Good morning. Καλημέρα σας. Έχουμε πολλές ψηφοφορίες που μας περιμένουν. Θα κάνουμε μια δοκιμή πρώτα. Ελπίζω να τα καταφέρουμε όλοι όσο γίνεται καλύτερα. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη πρώτα. Εγκρίνεται. Ναι. Ανακοινώσεις ότι έχουμε όλες τις γλώσσες για διερμηνία εκτός από μαλτέζικα και κροατικά. Σημείο 3. Παρουσίαση των διοργανικών διαπραγματεύσεων. Να έχετε να πείτε κάτι για την ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και πώς προχωράει ο τριμερής διάλογος, κύριε Κάσα. Όντως είμαστε στον τέταρτο και υπάρχουν κάποια προβλήματα με τη γονική άδεια. Από ό,τι φαίνεται, μπορεί να υπάρχει συμφωνία τελικά, όπως επίσης και για αυτούς που φροντίζουν. Πάντως η γονική άδεια είναι το πιο δύσκολο. Ελπίζουμε να υποχωρήσει το Συμβούλιο κάποια στιγμή. Θα το δούμε, θα το δούμε. Δεν ξέρω, δεν θέλω να σχολιάσω παραπάνω γι' αυτό. Οι συναντήσεις που γίνονται είναι πολύ τεχνικού χαρακτήρα. Πάντως η συνεργασία ήταν καλή μέχρι τώρα με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Θα δούμε λοιπόν τι θα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Τότε συνεχίζουμε και περνάμε στην ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις κάρτες σας, έτσι και αρχίζουμε να ψηφίζουμε με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Η Μαρία Ρενά είναι η συγγήτρια. Αρχίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 13. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 28. Όχι. Συγγνώμη, ναι, 25. 25 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την τροπολογία 25. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. Ίντα 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 29. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 15. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε για την 175 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος, απορρίφθηκε. Τροπολογία Τροπολογία 176. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κοντ 16. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 177. Με την Ρέγγι 21 που είναι ίδιες υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Συμβιβαστική 19. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 με την 196 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τις τροπολογίες 41 και 196 που ψηφίζουμε μαζί. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκαν. Συμβιβαστική 23. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κοντ 18 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 44, ψηφίστε, τέλος της προφορίας. Εγκρίθηκε με 21 ψήφους υπέρ. Τώρα, Τροπολογία 45. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Με 22 ψήφους κατά. Τροπολογία 46. Ψηφίστε ηλεκτρονικά. Τέλος, διακόπτη κάποιος. Α, τώρα τέλος και απορρίφθηκε με 23 ψήφους κατά. Τώρα. Ψηφίζουμε την τροπολογία 198. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 26, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 27, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 28, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 29, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 30 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 219 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε για τη 219 ηλεκτρονικά, μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της φοφορίας εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ. Κοντ 20 τώρα. Α, όχι, καταπίπτει, καταπίπτει, διορθώνει ο πρόεδρος. 221. Υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά 221. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε 51. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τροπολογία 223 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά 223. Ψηφίστε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Με 22 ψήφους υπέρ. 222 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 224 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε. 224 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. Με 26 ψήφους υπέρ. 225 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. 225 παρακαλώ ψηφίστε. Τέλος. Εν... Κρίθηκε. Με 23 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 31 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 32. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ίντα 25, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 236, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 238 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κόντου 23 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Κόντου 24, να ελέγξουμε, ωραία, για την 23 τότε, παρακαλώ ψηφίστε. Τέλος, εγκρίθηκε με μία ψηφοδιαφορά. Κόντι 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 231 έχει αποσυρθεί. 240. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 33 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 241 και 242 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 243 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 34 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 244 μαζί με την ή όχι. Όχι. Μόνη της. 244 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέγγι 35 υπέρ. Α, καταπίπτει αυτή. Ε, εντάξει, ναι. Επειδή 244 απορρίφθηκε, πρέπει να ψηφίσουμε τη ΡΕΚΙ 35. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ρέγγι 35. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. ...245 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 247 τώρα. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κόντι 25. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 57 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 248 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Κόντι 26 υπέρ, κόντι 26 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 46 and 60 Η 60 καταπίπτει, οπότε ψηφίζουμε το 249 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέγγι 36 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε Ρέγγι 36. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε με 30 ψήφους υπέρ. Τώρα, τροπολογία 250. <clears throat> Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Για να είμαστε σίγουροι, θα ψηφίσουμε τη ΡΕΚΙ 37. Ψηφίζουμε λοιπόν. Τέλος. Και εγκρίθηκε με 24 ψήφους υπέρ. Budget 9. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Νομίζω, αλλά θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Μπάτ 9. Τέλος. Εγκρίθηκε. Με 27. Δεν φαίνεται καλά από εδώ. Σηκώνετε τα χέρια σας παρακαλώ. 251 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. 251 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε. Με 22 ψήφους κατά. Ρέγγι 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Κόντι 27 υπέρ, κόντ 27, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την κόντ 27. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε με 22 ψήφους κατά. We vote on 253 τώρα μαζί με την 254. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκαν με 27 ψήφους υπέρ. 252 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 255 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κόντι 29 μαζί με την τροπολογία 67 που είναι ίδιες υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Ίντα 26 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Ίντα 26. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε. Με 23 ψήφους υπέρ. 256 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπατζ 10. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 257 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε. 257. Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ. Τέλος. Εγκρίθηκε. 26 ψήφι υπέρ. τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 259. Όχι. 260 και 261 ψηφίζουμε τώρα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Έγκρινεται. Κον 30, όχι. Ίντα, 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την ίντα 28. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε με δύο ψήφους διαφορά. Ρέγγι 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 34. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Εβδομήντα δύο τώρα, μαζί με την κόντ 31. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Απορρίφθηκε. ...263. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι 29. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 264 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι τα 30. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 266 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για το 266. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε με τρεις ψήφους διαφορά. Ρέτζι 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μπάτζ 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Μπάτζ 13. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπάτς 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μπάτς 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κον 32 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Κον 33. Θέλετε να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για την Κοντ 32. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ. Κον 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Κοντ 33. Ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 22 ψήφους υπέρ. 268 τώρα υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 269 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 271 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε 271 ηλεκτρονικά. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε με 28 ψήφους υπέρ. 270 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ρέτζιο 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 272 με την 78 μαζί και την κοντ 34 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 273 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 274 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ίντα 31 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κόντ 35 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε 35. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Τέλος. Εγκρίθηκε με 28 ψήφους υπέρ. Τροπολογία Ρέτζι 45. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε για την Ρέτζι 46. Τέλος, για τις 45 εγκρίθηκε με 27 ψήφους υπέρ. ...36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ρέντζε 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, εγκρίνεται, συγγνώμη. 275 υπέρ, κατά, αποχές, τα 32 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 276 απευθείας υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 47 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται με 27 ψήφους. Συμβαστική πρώτη. Ε, αιτιολογικές σκέψει. Δεν ψηφίζουμε την πρώτη συμβαστική. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική 91 μαζί με την ίντα 1 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική 2 κάνουμε έλεγχο πέρας απορρίφθηκε με 20 προς 17 πάμε στη Ρέτζη 2 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι τα δύο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Είναι τα δύο τα πέρας, απορρίφθηκε. Με μία ψήφου. Budget 1 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Πάμε στη συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Αιτιολογική 5. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ρέτζι 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 102 υπέρ, κατά, 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τα 6 υπέρ κατά αποχές κάνουμε έλεγχο για την Ίντα 6. Απορρίπτεται. Είναι τα 7 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Είναι τα 8 υπέρ, κατά, απόχέ, απορρίπτεται. Είναι τα 9 υπέρ, κατά, αποχέ απορρίπτεται. Πέρας, απορρίπτεται. 22 προ 17. Είναι τα 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 10 να κάνουμε έλεγχο. Πέρας, είναι τα 10. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Είναι τα 11. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Κοντ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ. 106 διορτώνει η πρόεδρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. τα 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. τα 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Είναι τα 14. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. 41 υπέρ, μία ψήφος κατά. <laughs> Ζητώ συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Δεν έβλεπα, λάθος γραμμή κοιτούσα. Τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Budget 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση της Budget 2. open and the is Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 6. Υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. 111 μαζί με την 112 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Όχι, ζητώ συγγνώμη, η ηλεκτρονική επαλήθευση. Μάλλον επαλήθευση, όχι ηλεκτρονική. Yes, Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας απορρίπτεται με 22 ψήφους κατά. 113. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 114. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Μαζί με την κοντ 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 115 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 118 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της 125 έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 14, έναρξη της ψηφοφορίας. Α, καταπίπτει. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος. Κοντ 6, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 16, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση είναι τα 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με τρεις ψήφους διαφορά. Κοντ 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είναι τα 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές η Ηλεκτρονική επαλήθευση 136. Έναρξη της ψηφοφορίας. 136. Λήξη της ψηφοφορίας. 33 ψήφοι υπέρ. Εγκρίνεται. Κοντ 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 137 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 142 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 143 υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Budget 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 15 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση της Ρέτζι 15. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 144 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται νομίζω. Ηλεκτρονική επαλήθευση. 144. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 29 ψήφους υπέρ. 145 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Την 22 δεν την ψηφίζουμε. Κοντ 10. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 146. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Budget 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της budget 6. Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Η 147 καταπίπτει, πάμε στην 148 και την 149 μαζί. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. 148 και 149. Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνονται με 24 ψηφούς υπέρ. Η 150 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε λοιπόν το σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη της ψηφοφορίας για την τελική ψηφοφορία. Λήξη της τελικής ψηφοφορίας και εγκρίνεται η έκθεση με 42 ψήφους υπέρ, μία ψήφο κατά. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια για όλη τη δουλειά που έχει κάνει.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 Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 23 ψήφους κατά. Τροπολογία 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 114 ζητάει κάποιος. Ελέγχουμε λοιπόν. Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με διαφορά δύο ψήφων. 115 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 117 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 120 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 125 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 125 έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. 126 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση πάλι της 126 έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Με 24 ψήφους κατά. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 131 υπέρ. Κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της 131. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 23 ψήφους κατά. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Συμβαστική 12. Έναρξη της ψηφοφορίας. Is now on 12. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Amendment 134. 134 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 135 και 136 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση 144. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Κάποιος ζητά ηλεκτρονική επαλήθευση. 146. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 23 ψήφους κατά. 196 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 148 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 148. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 149 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 150 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 151 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 169, καταπίπτει. Συμβαστική 16, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 156 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά, Αποχέ εγκρίνεται. 160 υπέρ, κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 160. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 22 ψήφους κατά. 161 υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 162. 162. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 163. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 170. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 173. Μαζί με την 174. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 175. 175 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της συμβαστικής 21, άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Συμβαστική 21 εγκρίνεται με 23 ψήφους υπέρ. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 186 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ. Κατά. Αποχές Ηλεκτρονική επαλήθευση 187. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με δύο ψήφους διαφορά. 188. Υπέρ. 188. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 190 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 δεν την ψηφίζουμε. 193 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 195 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 δεν την ψηφίζουμε. 199 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση της 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Τροπολογία 22. Απορρίπτεται. Τροπολογία 200. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 202. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ, κατά, αποχές Ελέγχουμε για 24, 204. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 προς 19. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. <laughs> Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Πέρας για την 25. Απορρίπτεται με 24 ψήφους. 210. Όχι. Α, 206 του κυρίου Ντέτσχεν υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 207 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 208 υπέρ, κατά, αποχές, 209 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 210 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 211 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Ε, να ελέγξουμε για 211. Πέρα. Εγκρίθηκε 212 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 213 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 215 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 216 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 49 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. 227 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 230 και 31 ταυτόσημες μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 230 και 31. 200 η συμβαστική 26 υπέρ. Α, δεν ψηφίζουμε. Συμβαστική 27 δεν ψηφίζουμε. 233 235 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 28 δεν ψηφίζουμε συμβαστική 29 υπέρ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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. 252 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 250 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 253 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 255 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 39 39 στη σελίδα 15 για μένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα. 273. 274 και 275. Μαζί, ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 276 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 277 και 278 ταυτόσιμες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 282 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα τα παραρτήματα. 283 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 284 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 285 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 286 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 287 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 288 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 289 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 290 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 289. Τι 290 θέλετε να ελέγξουμε ελέγχουμε, άρχεται η ψηφοφορία. <clears throat> Πέρας. Απορρίφθηκε. ...291 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 292 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 293 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 294 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 295 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 296 υπέρ. Κατά. Αποχές. Για να ελέγξουμε. 296 έρχεται η ψηφοφορία. 296 πέρας απορρίπτεται 23 ψήφοι κατά 297 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 298 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 299 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Καλά, να σε ελέγξουμε τα 299. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρα. Ναι, εγκρίθηκε με 32 ψήφου. 300 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 301 υπέρ, κατά, απόχέ απορρίπτεται. 300... Θέλετε έλεγχο για την 301. Απορρίφθηκε 301. 302 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 303 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 304 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 305 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 306 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 307 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 308 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 309 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 310 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, απορρίπτεται, συγγνώμη. 310 πέρας εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Πέρας. Απορρίφθηκε με μία ψηφοδιαφορά. 311 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 315 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 316 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 318 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Κατευθείαν στις ιδεολογικές σκέψεις τώρα. Με τη σκέψη παριθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Με τη 2 υπέρ, κατά, αποχές, έλεγχος. Έλεγχος για την αιτιολογική 2. Πέρας. Εγκρίθηκε. 22 ψήφι υπέρ. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική υπαριθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 62 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 63 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 64 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. Έλεγχος. «64 άρχεται ψηφοφορία, πέρας, απορρίπτεται. 23 ψήφοι κατά. 65 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, ε, εγκρίνεται. Αιτιολογική 12, 67 τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Καταπίπτει 70, όχι 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 72 υπέρ, κατά, αποχές. Εγώ νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά να το ελέγξουμε καλύτερα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 72, πέρας και εγκρίθηκε με 20 ψήφους. «73. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 75. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπεται 77 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 78 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79, 80 και 81 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνονται. 82 υπέρ. Α, καταπίπτουν και 83. Πρώτο τμήμα της 84, The ESF Plus, Part Under Management. Πρέπει να ε, ψηφιστεί ως προσθήκη στην Συμβαστική 5, υπέρ. Κατά αποχές θα έλεγα να ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Στο πρώτο τμήμα. Απορρίφθηκε με 24 ψήφους κατά. 86. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 87 και 88 μαζί, ταυτόσιμες, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. 89 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε την 89 ε, ε, Πέρας. Εγκρίθηκε με 40 ψήφου και μία κατά. Αλλά κανεί δεν σήκωνε το χέρι του. 90. Υπέρ. Κατά. απόχέ. Εγκρίνεται. 91 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Πρέπει να ελέγξουμε για την 91. Άρχεται η ψηφοφορία. Τώρα τελείωσε. Εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ. Πρώτο τμήμα, το ESF SYN και η κοινή διαχείριση, το Set Management. Προσθήκη στη συμβαστική 6. Υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 97 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. 99 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 100 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Αιτιολογική 60. 102. Δεύτερο τμήμα. Το ESF συν και η κοινή διαχείριση. Είναι ε, η προσθήκη στο 7. υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 104 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Συμβαστική 8. Δεν θα ψηφιστεί. 105. Το πρώτο τμήμα το ESF και η κοινή διαχείριση θα είναι προσθήκη στη συμβαστική 8. Υπέρ. Κατά. Ξανά. Για να είναι σαφές. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 109 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 110. Να κάνουμε έλεγχο για την 109. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Α, μάλιστα. Απορρίφθηκε με ισοψηφία. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίφθηκε. 111 υπέρ τα αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία ονομαστική. Άρχεται. Τώρα τελείωσε. Εγκρίθηκε. Με μικρή διαφορά. 22 προς 18 και μία αποχή. Ευχαριστούμε πολύ για όλη σας τη σκληρή δουλειά. Then you have the new... Περνάμε στο επόμενο θέμα, δημιουργία μιας ευρωπαϊκής λειτουργίας σταθεροποίησης επενδύσεων. Ο επόμενος κατάλογος ψηφοφοριών. Άρθρο 1, παράγραφος 2, τροπολογία 91. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 106 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Υπάρχει μια προφορική τροποποίηση του εισηγητή. Ένα μεγάλο συμμετρικό σοκ. Ή μια σημαντική αλλαγή κλπ. Λοιπόν, αυτό το δεύτερο κομμάτι διαγράφεται. Το or significant downturn υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Ωραία. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν για την τροπολογία 113. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. απορρίφθηκε με 28 ψήφους κατά. Τώρα, τροπολογία 25 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 με την ίδια τροπολογία, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 27 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 114 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 28 με την προφορική τροποποίηση υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Θέλετε να ελέγξουμε. Καλώς ελέγχουμε για την τροπολογία 28. Μπορείτε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά. Τέλος. Όντως εγκρίθηκε με 23 ψήφους υπέρ.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 115 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε για την 37 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος ψηφοφορίας. Και εγκρίθηκε με 22 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 38. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 17. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 16. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 41. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 121 μαζί με την 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Τώρα, αιτιολογική σκέψη, συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 45 υπέρ, κατά, αποχές. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 45. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίφθηκε. 23 ψήφους κατά. Απορρίφθηκε. Και συνεχίζουμε. Τροπολογία 46. Υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε για την 46 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος, απορρίφθηκε με 24 ψήφους κατά. Συμβαστική τροπολογία 2. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ, κατά. Θα ελέγξουμε τη συμβαστική 4 ηλεκτρονικά για σιγουριά. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε 24 ψήφοι υπέρ. Τροπολογία 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 61 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 62 υπέρ, κατά, δεν είμαι σίγουρη να ελέγξουμε καλύτερα για την 62 ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος. Απορρίφθηκε με 24 ψήφους κατά. Συμβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 66. Τώρα η 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα 67 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 68 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 69 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 70 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 71 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Ωραία, 71. Ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε 24 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 10. Υπέρ. Κατά. Να ελέγξουμε ηλεκτρονικά για τη 10. Ψηφίστε. Τέλος. Εγκρίθηκε 22 ψήφι υπέρ. 30 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 81 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 82 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 83 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 85 δεύτερο τμήμα ως προσθήκη στη συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε άμα θέλετε για το δεύτερο τμήμα Δεύτερο τμήμα. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίφθηκε. Τώρα τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 12. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος. Εγκρίθηκε. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 9 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία 9. Μπορείτε να ψηφίσετε. Τέλος της φοφορίας. Εγκρίθηκε 21 ψήφι υπέρ. Οπότε τώρα ψηφίζουμε με ονομαστική ψηφοφορία την τροποποιημένη, το τροποποιημένο κείμενο. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος, εγκρίθηκε 26 ψηφί υπέρ, 3 κατά και 11 αποχές. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτή την ψηφοφορία και ευχαριστώ και την εισηγήτρια. Τον εισηγητή, συγγνώμη, τον κύριο Σομπού. Θα ψηφίσουμε τώρα το σχέδιο γνωμοδότησης για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών. Το e ΕΝΕΦ ζήτησε ονομαστικές ψηφοφορίες, ε, έχει αποσύρει όμως πάλι το αίτημα. Και ξεκινάμε από την τροπολογία 4, υπέρ. Κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση. 4, τροπολογία 4, έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται με, 25, με 21 ψήφους κατά. Τροπολογία 5 υπέρ. Η ηλεκτρονική επαλήθευση και τις 5. Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, τροπολογία 5. Απορρίπτεται. Άρθρο 1, παραγραφός 1, σημείο 4, τροπολογία 26. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 26. Λήξη της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Τροπολογία 6. Έναρξη της ψηφοφορίας για την τροπολογία 6. Vote is now Λήξη της ψηφοφορίας εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. 20 ψήφους δηλαδή. Τροπολογία 7. Υπέρ. Εκτός μικροφώνου δεν ακούμε. Do you want us to repeat? Yes, thank you. Θέλετε να επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Ναι, παρακαλώ. Ο κύριος Ανωνάτο.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 We will repeat uh, the vote on amendment Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 6. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 7. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Έχουν αποσυρθεί όλα τα αιτήματα του ΕΝΕΦ e για ονομαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε πάλι. Τροπολογία 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 32 καταπίπτει. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά η ηλεκτρονική επαλήθευση, συμβιβαστική 7. Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. Η 35 καταπίπτει. 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 37 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση της 37. Έναρξης ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Τροπολογία 37. Απορρίπτεται με 23 ψήφους κατά. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 38. Για να είμαστε βέβαιοι. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με μία ψήφο διαφορά. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Η ηλεκτρονική επαλήθευση της 10. And the vote is open and now... Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 22 ψήφους κατά. Τροπολογία 11. Ε, ηλεκτρονικά θα ψηφίσουμε. Έναρξη της ψηφοφορίας για την τροπολογία 11. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με δύο ψήφους διαφορά. Τροπολογία 12. Έναρξη της ψηφοφορίας. Τροπολογία 12. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 19 ψήφους υπέρ. Τροπολογία 13. Έναρξη της ψηφοφορίας. And the vote is now closed on a... Λήξη της ψηφοφορίας για την τροπολογία 13. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. 43. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 8. Υπέρ, κατά, αποχές, ηλεκτρονική επαλήθευση. Έναρξη της ψηφοφορίας, συμβαστική τροπολογία 8, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με 25 ψήφους υπέρ. 14 υπέρ. Κατά. Η ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογία 14, έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με 34 ψήφους υπέρ. 47. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 1, υπέρ. Κατά, αποχές Εγκρίνεται νομίζω. Ηλεκτρονική επαλήθευση, συμβαστική 1. Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ. Ε, αιτιολογική σκέψη 6 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 2. Έναρξη της ψηφοφορίας. Λήξη της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 21 ψήφους κατά. 17 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ. Κατά ηλεκτρονική επαλήθευση, τροπολογία 3. Έναρξη της ψηφοφορίας, τροπολογία 3. Λήξη της ψηφοφορίας, εγκρίνεται με 28 ψήφους υπέρ. Συμβαστική 2. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση, συμβαστική 2. Έναρξη της ψηφοφορίας, λήξη της ψηφοφορίας και εγκρίνεται με 26 ψήφους υπέρ. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε το σύνολο του σχεδίου γνωμοδότησης όπως τροποποιήθηκε. Έναρξη της ψηφοφορίας. Τελική ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ, 17 ψήφους κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια στην κυρία Ριμπέιρο. για τη δουλειά της πάνω στη γνωμοδότηση αυτή. Η επόμενη συνεδρία θα πραγματοποιηθεί 3 Δεκεμβρίου. Δεν είχαμε χρόνο για συζήτηση σήμερα, μόνο τις ψηφοφορίες ε, κάναμε. Θα σας δω λοιπόν τότε. Αργά το απόγευμα θα συνεδριάσουμε 4 με 6.30. Θα τα πούμε το Δεκέμβριο.